Ε, μη συμβατά με αυτά του ε, Ευρωβουλευτή. Τρίτη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ενημέρω... Ε, διαβίβασαν στο Κοινοβούλιο την... το αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της κυρίας Μαρή Λεπέν. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Τέταρτη ανακοίνωση. Σας ανακοινώνω από την ομάδα ALDE και από την